για το 2015. Δίνω το λόγο εκ μέρους του Συμβουλίου στον κύριο Κόνης. Thank you Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι γίναμε μάρτυρες ε, σημαντικής πρόοδου στη σχέση μας με τη Σερβία πέρυσι. Με επιστέγασμα την έναρξη των πρώτων δύο κεφαλαίων διαπραγμάτευσης. Έτσι ε, έχει πάρει σάρκα και οστά η δεξιακή διαδικασία και χαράχθηκε η μελλοντική πορεία. Κάτι που είναι αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών και της δέσμευσής μας. Πολύ θετικά μαντάτα δηλαδή. Και μάλιστα το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ε, υποβολή εκ μέρου Σερβίας του σχεδίου δράσης για το κράτος δικαίου. Και περιμένουμε φυσικά την πιστή εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης και ένα μικρό αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τη νέα προσέγγιση, ε, περιμένουμε το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24 που θα τεθούν σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Η πρόοδο στα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να γίνει παραλλήλου με τις συνολικές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των κεφαλαίων που άνοιξαν ε, το καλοκαίρι, το 35 που αφορά την εξομάλυση των σχέσεων ε, Πρίστινα Βελιγραδίου έχει κεφαλαιώδη σημασία και μάλιστα η συμφωνή ορόσημο που έγιναν τον Αύγουστο για τη, για τη διευκόλυνση του διαλόγου συνιστούν σημαντική ε, επιτυχία. Πολιτικά η κατάσταση δεν ήταν καθόλου εύκολη και θα ρίναμε τη Σερβία να συνεχίσει την επικοδομητική τη ε, προσπάθεια εφαρμόζοντα το δικό τη θύμα των συμφωνηθέντων. Έχουμε παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς ε, τι εξελίξει αυτέ και η εξομάλυνση στο σχέση με το 25 θα πρέπει να συνοδεύεται ε, με την πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας. Η Σερβία έχει διαδραματίσει πολύ θετικό και επικοδομητικό ρόλο στη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης από την οποία επηρεάστηκε πολύ σοβαρά. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίσιμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα στηρίξουμε τη τεχνικά και χρηματοοικονομικά τη Σερβία και στο τομέα αυτό. Το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την ε, ιδιαίτερη επικοδομητική δέσμευση της Σερβίας στην περιφερειακή συνεργασία και την ενίσχυση των αγαθών σχέσεων γειτονία. Μάλιστα, ο ρόλο τη Σερβία θα είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ευρύτερη σταθερότητα τη περιοχή. Είναι και σημαντικό εταίρωση τη εξωτερική μα πολιτική. Και τη συγχαίρουμε για την επιτυχή προεδρία τη ΟΑΣΕ που είχε αναλάβει το 2015. Επίση, από κοινού θα αντιμετωπίσουμε τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κυρίως ε, στη γειτονία μας. Γι' αυτό και θα θέλαμε η Σερβία σταδιακά να ευθυγραμμιστεί με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μια φιλοευρωπαϊκή Σερβία ανήκει στο κοινό μα όραμα. Γενικώ μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ενταξιακή μα πολιτική προ τη Σερβία απέδωσε καρπού πέρυσι. Βέβαια, περιμένουμε διάφορα από τη Σερβία. Για παράδειγμα, ενίσχυση των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και πιστή εκτέλεσή του, ιδιαίτερα στη δικαστική μεταρρύθμιση, την πάταξη τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο, καθώ και την εξασφάλιση τη ελευθεροτυπία και τη ελευθερία μέσων μαζική ενημέρωση. Επίση, προβλέπουμε περαιτέρω πρόοδο στην εφαρμογή των συμφωνιών με το Κωσυφοπαίδιο. Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστούμε ότι οι πρόορε νομοθετικέ βουλευτικέ εκλογέ στη Σερβία δεν θα επιβραδύνουν αυτή τη διαδικασία. Επίση, θα πρέπει οι βουλευτικέ αυτέ εκλογέ να γίνουν ε, σε συμφωνία με τι διεθνεί προδιαγραφέ και προβλέπουμε στο περαιτέρω άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με τη Σερβία κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ο Επίτροπος Χάν λαμβάνει το λόγο τώρα εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Κύριε ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω τον, τον ε, Υπουργό Ιωξίμοβιτς και την αντιπροσωπεία που τον συνοδεύει. Θέλω ταυτόχρονα να συγχαρώ τον Ντέβιτ Μακάλιστρο για το ψήφισμά του για την έκθεση πρόοδου 2015 για τη Σερβία. Πρόκειται για μια αξιολόγηση ισορροπημένη, καλή, της πρόοδου της Σερβίας στην ε, στα πλαίσια που έχει ορίσει και η δική μας έκθεση πρόοδου. Έχει προχωρήσει στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Σορβίας. Συμμερίζομαι την θέση ότι έχει επιτύχει πολλά προς τον στρατηγικό της στόχο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πραγματοποιήσει συγκεκριμένες προόδους για ε, την υλοποίηση ενός φιλόδοξου οικονομικού και τερθωτικού προγράμματος. Είναι προσιλωμένη στη βελτίωση των περιφερειακών και δημερών δεσμών σε συνθήκες ε, καλής γειτονίας. Έχει πραγματοποιήσει προόδους για τη μεταρρύθμιση του κράτους, των κρατικών δομών και την ενίσχυση του κράτους δικαίου με την υιοθέτηση διατάξεων και την εξομάλυνση των σχεσιών της με το κοσφοπέδιο κύριας ε, σημασία ήταν οι συμφωνίες του περασμένου Αυγούστου. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τον ε, πολύ ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο η Σερβία και οι Σέρβοι πολίτες αντιμετωπίζουν το μεγάλο αριθμό και τις προσφυγικές ροές. Όλα αυτά είναι, δείχνουν σεβασμό των ε, κύριων αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των δύο πρώτων διαπραγματευτικών κεφαλαίων 32 και 35 συγκεκριμένα που άνοιξαν το Δεκέμβριο του 2015 σε ένδειξη αναγνώριση αυτών των προσπαθειών. Τώρα πρέπει λοιπόν να οικοδομήσει πάνω σε αυτήν την πρόοδο η Σερβία να προχωρήσει αποφασιστικά στις μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στο χώρο της δικαιοσύνης, δικαστικής εξουσίας, της καταπολέμησης διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ελευθερίας της έκφρασης, των κρατικών δομών, την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων και της οικονομίας ταυτόχρονα. Η Σερβία πρέπει να συνεχίσει την επικοδομητική της προσέγγιση και την πρόοδό της για την εξομάλυνση των σχέσεων της με το κοσφοπέδιο. Παράλληλα, με τη διαδικασία προσχώρησης θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό για να υπάρξει μια πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων όπως στοχεύει το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Προσβλέπω επίσης στο επόμενο βήμα που είναι ε, το άνοιγμα των ε, κεφαλαίων 23 και 24 που αφορούν το κράτος δικαίου και όπως και ο εισηγητής κ. Μακάλιστερ ελπίζω ότι αυτό θα καταστεί δυνατόν κατά το πρώτο εξάμεινο του 2016 φυσικά πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες της Σερβίας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και εν προκειμένου καλώς ορίζω το πρόγραμμα δράσης ε, που αναφέρεται ειδικά στις μειονότητες και που δημοσίευσε σήμερα στις Βρυξέλλες η Σερβία. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και μια ταχύτατη πορεία προς τα επόμενα βήματα συμφωνίας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην επιβαρύνουμε με επιπλέον ε, απαιτήσει που δεν απαιτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή το ε, διαπραγματευτικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να μην παρεμποδίσουν την όλη διαδικασία προσχώρησης δημιουργείς ε, διαφορές και εν τέλει καταγράφουμε την ανακοίνωση από πλευρά της κυβέρνησης Σερβίας που πρόκειται να διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές και ελπίζουμε ότι τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και μετά την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρνησης θα παραμείνει προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό τη ε, θεματολόγιο και την εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσμοπέδιο της Σερβία. Κυρίε και κύριοι, η Επιτροπή είναι προσιλωμένη στο έργο τη της καθοδήγησης και τη υποστήριξη τη Σερβία σε αυτή την πορεία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω πω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται στο ίδιο μήκος κύματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. πρώτο ομιλητή εκ μέρου των πολιτικών, πολιτικών ομάδων, εκ μέρου του ο Μακαλίστερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πριν τα Χριστούγεννα η, Σέρβια, η Σερβία έκανε ένα τεράστιο βήμα πρόοδου για την προσχώρηση στην Ένωση. Δύο χρόνια μετά από την ανάγκη των συνομιλιών προσχώρηση με την Ένωση και λίγου μήνε μετά την νέα συμφωνία με το Κωσυφοπαίδιο, άνοιξαν τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση. Η κυβέρνηση και ο, ο κ. ο οποίος είναι σήμερα εδώ, δείχνουν τη δέσμευσή τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θα ήθελα να τονίσω τέσσερα κυρία σημεία καταρχάς στο ψήφισμα Πρώτα το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. Όταν αυτό εφαρμόζεται είναι καλό για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για την οικονομία, για την κυβέρνηση. Η Σερβία λοιπόν θα πρέπει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά και το δικαστικό σώμα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Δεύτερον, η δημοκρατία. Το πίσω αυτό τονίζει τη σημασία του ενεργού ρόλου του Κοινοβουλίου και την εργό και επικοδομητική συμμετοχή δυνάμεων που είναι τόσο σημαντικές για την κοινωνία της Σερβίας. Τρίτον, ελευθερία ΜΜΕ. Ελευθερία εκφρασής είναι ένας πυλώνας δημοκρατίας που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υιοθέτηση νομοθεσίας. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθεί και ένα πλαίσιο για ανεξάρτητα ΜΜΕ. Και τέλο, τέταρτο, περιφερειακή συνεργασία. Σχέση καλή γειτονία νομίζω αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη διαδικασία προ την Ένωση. Η δέσμευση τη Σερβία και ο ρόλο τη στην προώθηση τη περιφερειακή συνεργασία και η συμφιλίωση στα Βαλκάνια είναι ευπρόσδεκτο. Η πιο πρόσφατη συμφωνία στα πλαίσια αυτού του διαλόγου νομίζω ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου για την ομαλοποίηση, για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσμοπεδίου και Σερβίας και τα δύο τώρα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις συμφωνίες. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω προς την Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου θεωρώ ότι τα κεφάλαια 23-24 θα πρέπει να ανοίξουν ταχύτερο δυνατό ώστε να βοηθήσουμε την Σερβία όσο γίνεται στον δρόμο προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τάνια Φαγιών έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόοδος που έχει επιτελέσει τα τελευταία χρόνια η Σερβία ακορυφώθηκε με το άνοιγμα δύο κεφαλαίων διαπραγμάτευση ε, για το δημοσιονομικό έλεγχο και την εξομάλυση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας. Είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδου, αλλά αναμένονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Χαιρετίζουμε το ψήφισμα και απευθύνουμε και εμείς έκκληση για το άνοιγμα κεφαλαίων, των κεφαλαίων 23 και 24 το συντομότερο δυνατό γιατί θα έχουν κέρια σημασία για τη μεταρρύθμιση της σερβικής κοινωνίας. Με βάση τη δική μας εμπειρία στη Σλοβενία, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε αμύωτο το ρυθμό και τη δυναμική των διαπραγματεύσεων. Και ελπίζω ότι οι πρόορες βουλευτικές εκλογές δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον ταχύ ρυθμό μεταρρυθμίσεων στη Σερβία. Η Σερβία, χρειάζεται, η Σερβία χρειάζεται μια σαφή ε, και συσπηρωμένη θέση σε ό,τι αφορά το, την ενταξιακή της πορεία. Χρειάζεται εμπειρογνώμονες ε, με ενέργεια και ενθουσιασμό για να υλοποιήσει τους στόχους της για μια ισχυρή Σερβία, σύγχρονη, οικονομικά ευημερούσα με σημαντικό ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Σερβία δεν χρειάζεται ούτε πολιτικοποίηση, ούτε εγωιστικά πολιτικά συμφέροντα ε, που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερισχύουν των κοινωνικών συμφερόντων. Ποιο είναι υπεύθυνο για την κατάσταση τα μέσα μαζική ενημέρωση τη Σερβία. Ω πρώην δημοσιογράφο, θα ήθελα να αναφέρω τα επεισόδια του τέλου του έτου και τι ε, απρεπεί ε, δηλώσει ε, του Υπουργού για τις γυναίκες δημοσιογράφους που ήταν έτοιμες ε, να γονατίσουν. Αυτό έριξε λάδι στη φωτιά σε ό,τι αφορά την κατάσταση το μέσο μαζικής ενημέρωσης ε, στη Σερβία και σίγουρα δεν είναι αυτή η πορεία που θα ήθελα να δω τη Σερβία να ακολουθεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και στους νέους Σέρβους, στη νεολαία της Σερβίας και να αποτρέψουμε τη μαζική τους έξοδο από την πατρίδα τους. Σε αυτό το θέμα θα αφιερώσουμε όλοι μας την προσοχή, γιατί αν χάσουν οι νέοι την ελπίδα τους στο σερβικό μέλλον, σίγουρα δεν θα είναι καλό σημάδι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Στάνοκ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω συνεργαστεί με τον Ντέβιτ Μακάλιστερ και επί την αίσθηση του Μαυροβουνίου. Θέλω να τον συγχαρώ λοιπόν. Η Σερβία βρίσκεται σε πρώιμα βήματα τη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μόλι ολοκληρώσει τη διαδικασία τη επισκόπηση τη ε, νομοθεσία ε, το 2015 το Μάιο, αλλά σημειώνονται σημαντικέ προόδειε προ το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι προ τη δυνατότητα τη Σερβία να συνεχίσει αυτή την πορεία παρά τις ε, πιέσεις ει ε, προσφυγικής κρίσης. Βέβαια τη βοηθάει το γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις και ο διάλογος με το κοσμοπέδιο. Οι σχέσεις Μαυροβουνίου-Σερβίας παραμένουν ισχυρές και εξελίσσονται. Υπάρχει μια ε, συμφωνία συνεργασία εν εξελίξη και μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο και για την καταπολέμηση της ε, διασυνοριακής εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος. Τα κεφάλαια 23-24 συμφωνώ με τον David πρέπει να ανοίξουν ταχύτερο δυνατό και σε σχέση με τα δεδομένα ασφάλειας έχουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα με την εφαρμογή του 2015 φυσταμένων συμφωνιών που στόχο έχουν να βελτιώσουν και στο θέμα των τηλεπικοινωνιών τις ε, τα τέλη περιαγωγής αλλά και να παρακολουθήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Το Βελιγράδι πιστεύω ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί περισσότερο στι στις του κεφαλαίου 31 σε σχέση με την ΚΕΠΑ και κυρίως τι κυρώσει προς τη Ρωσία. Αυτή είναι η σύστασή μου. Είναι κλειδί για τα Βαλκάνια η Σερβία. Είναι ένα κομμάτι τη σταθεροποίηση ολόκληρη τη περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά δηλώνω ότι η ομάδα μας υποστηρίζει τη Σερβία και τις προσπάθειές της για την τήρηση των προϋποθέσεων όσον αφορά την ευθυγράμμιση με τους κανόνες που οδηγούν στην προχώρηση στην Ένωση. Ευχαριστώ τον κύριο Μακάλιστερ, τον εισηγητή τη θαυμάσια δουλειά του και το έγγραφο, όπως επίσης και για τη συνεργασία με τους κύριους εισηγητές. Να μην ξεχνάμε ότι κάθε χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που θέλει να προσχωρήσει στην Ένωση θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή προοπτική. Ξεκινάμε από την αρχή ότι το κράτος δικαίου αποτελεί την βάση των πολιτικών διεύρυνσης και συνειδητοποιούμε ότι η Σερβία ήδη έχει κάνει πάρα πολλά σε σχέση με την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το ότι η πολιτική είναι υπερβολικά παρούσα στα ΜΜΕ. Αυτές λοιπόν οι πολιτικές είναι ιδιαίτερα ενσυχητικές όσον αφορά δηλαδή το πεδίο των ΜΜΕ. Θα πρέπει η μάχη για την ελευθερία των ΜΠΕ να μην περιοριστεί μόνο στην προώθηση του ισχυόντος κατεστημένου. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει και αυτή να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατικής αυτής διαδικασίας και όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από την εξουσία για να υπερισχύσει. Η Σερβία λοιπόν θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες εξωτερική ασφάλεια και τη εξωτερική πολιτική, γιατί η Σερβία δεν έχει άλλε αναλλακτικέ λύσει. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρόοδο όσον αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων με το Κωσυφοπέδιο αλλά θεωρώ ότι η πρόοδο στη συνολική θα εξαρτηθεί και από του δύο. Πρέπει λοιπόν η ενίσχυση τη συνεργασία στην Σερβία να είναι περιεκτική και αυτή ακριβώ θα πρέπει να είναι κατά τη συγκέντρωση τη πολιτική εξουσία. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε γαλάζια κάρτα τον κύριο Φρουντσούλικα. Μάλιστα, έχετε το λόγο κύριε Φροντσούλικα. Α, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώ εδώ ως ε, φίλος της Σερβίας. Ερωτώ όμως, γνωρίζουμε ότι η Σερβία θα πρέπει να επιφέρει πολλές βελτιώσεις ό,τι αφορά το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια των εθνικών μειονοτήτων. Έχει ακόμη δρόμο να κάνει. Και μερικέ φορές ε, η σερβική κυβέρνηση, οι μέλη τη σερβική κυβέρνηση έχουν κάπως αντιευρωπαϊκή ρητορική. Δεν πρέπει να απόσχει από τέτοιε δηλώσει ε, η σερβική κυβέρνηση και να μην προσπαθεί να χειραγωγεί και το κοινό στα θέματα αυτά. Ποια είναι η γνώμη σας. Ο κύριος Βάγκλ. Είπα στην ομιλία μου ότι η Σερβία θα πρέπει να είναι πολύ σαφής και να ταχθεί υπέρ της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε χρήσιμο ούτε επικοδομητικό για την ίδια και για την ενταξιακή διαδικασία να φλερτάρει η χώρα με την Ρωσία. Δεν είναι αυτή η εναλλακτική για τη Σερβία. Ο κύριος Χατζηγεωργίου έχει το λόγο. Συγγνώμη. που δεν προφέρω σωστά το όνομά σα. Συνάδελφοι, οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων έχουν περάσει μέσα από πάρα πολλέ δυσκολίε, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90, μέσα από πολλού πολέμου και πάρα πολύ αίμα. Σήμερα όμω βρισκόμαστε σε μια νέα φάση, στην οποία καταβάλλεται έντονη προσπάθεια να επιληθούν ζητήματα, όχι με τα όπλα αυτή τη φορά, αλλά μέσα από το διάλογο και τη θέληση τη συνεργασία η ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει να σταθεί συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση στο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ βελιγραδίου και πρίστινας για εξέβρεση πολιτικής λύσης στο ζήτημα του κωσυφοπεδίου. δεν επιτρέπεται κατά την άποψή μας η ευρωπαϊκή ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερα αυτό το κοινοβούλιο να υποδαβλίζει αυτή την προσπάθεια και αυτό το διάλογο. η οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα του διαλόγου μεταξύ πρίστινας και σερβίας. υποστηρίζουμε ως ομάδα την ενταξιακή πορεία της σερβίας ωστόσο διαφωνούμε με τη στάση της ένωσης που εκφράζεται μέσα στην έκθεση και παρεμβαίνει στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής ε, της σερβίας αλλά και στην επιβολή οικονομικών μοντέλων που αποδεδειγμένα έχουν επηρεάσει σε τόσο αρνητικό βαθμό τους λαούς της ευρώπης. ας εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας να στηρίξουμε τη χώρα στις προσπάθειες που κάνει για αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχει για εμβάθυνση του κράτους δικαίου αντιμετώπιση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και των προσφυγικών ροών που τον τελευταίο καιρό φτάνουν στη χώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Σόλτες είναι ο επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ για την έκθεσή του. Ξέρετε η έκθεση και θέλω να ευχαριστώ και όλους τους συνεισηγητές και οδησηγητές για τη συνεργασία τους το ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στην πρόοδο κατά το 2015 της Σερβίας και την έκθεση είναι πληρέστατο. Περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά θέματα. Η Σερβία πιστεύω έχει πραγματοποιήσει μεγάλες προόδους, κυρίως το αποδεικνύει το άνοιγμα των δύο διαπραγματευτικών κεφαλαίων και φαντάζομαι ότι και η κυβέρνηση Σερβίας θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τους ίδιους ρυθμούς και τη δυναμική που έχει μέχρι τώρα επιδείξει είναι ωστόσο απολύτως απαραίτητο να παραμείνει σημαντικός παράγων στις σχέσεις στα δυτικά, μεταξύ των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων η Σερβία. Με καλές σχέσεις μεταξύ των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής μπορεί να προοδεύσει όλη η περιοχή. Ο κ. Μακάλιστερ υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία του κράτους δικαίου, το οποίο έχει απήχηση στα πάντα, το, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και σειρά άλλων στοιχείων. Όπου πάντα βεβαίως μπορεί κανείς να επιφέρει υπέραιτερα βελτιώσεις. Πάντα χωρούν βελτιώσεις. Οι σχέσεις με τον μη κυβερνητικό τομέα βελτιώνονται βεβαίως, αλλά πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να μπορέσει να συμμετάσχει στο του επίπεδο στη διαδικασία των κλεισλήψεων των αποφάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέσα μαζική ενημέρωση, ε, τον έλεγχό του, την κατάσταση εργασίας, επιτέλεση του έργου των δημοσιογράφων ε, θα ήθελα να σημειώσω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα οι δημοσιογράφοι να κάνουν τη δουλειά τους όπως την εννοούν έστω και αν αυτό δεν ε, είναι πάντα ευχάριστο για τις αρχές. Επίσης η Σερβία έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της αντιμετώπισης των, ε, της ολοκλήρωσης και πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε το δημοσίευμα στη Βρετανία για τη συμμετοχή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε οι Βρετανοί δεν θα ψηφίζουν μόνο για τι σχέσει μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τι φιλοδοξίε στην νεοπικιοκρατικές τη Ένωση υπό το φω τη τωρινή κρίση, Χώρε όπω η Ιδία, η Γερμανία, η Βρετανία νομίζω ότι ε, βρέθηκαν σε μια κατάσταση που πίεσε τη Σερβία και γι' αυτό ακριβώ θέλουμε να θεωρήσουμε τη στάση μα. Κυρία Πρόεδρε, έχει η Ένωση προτείνει λύσει για την τωρινή κρίση του προσφυγικού, για τα σύνορα. Αυτή η μάσα ανθρώπων, αυτή η μάζα ανθρώπων νομίζω ότι ε, θεωρείται ως κάτι το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση. Έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και νομίζω ότι αυτό ακριβώς δικαιολογεί την θέση του κυρίου Κάμερον για επαναδιπραγμάτευση της παρουσίας μας στην Ένωση και νομίζω ότι ε, ε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Κυρία Πρόεδρε, όσο είμαστε στην Ένωση το μέλλον της Βρετανίας δεν είναι σαφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαφχάουζερ, επόμενος ομιλητής. μισή λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Σερβία σίγουρα έχει ε, βλέψεις και ενταξιακή πορεία. Και ακόμη και χρειάζεται κάποιες επιπλέον προσπάθειες ό,τι αφορά την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Γιατί αν η έκθεση αυτή επιδιώκει την ισορροπία γιατί να, αποκα... να αποκρύψουμε τις ε, δράσεις εις βάρος ε, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των ε, ορθόδοξων σερβικών θρησκευτικών μειονοτήτων που έγιναν στο Πέδιο, που είναι μαφιόζικο κράτος. Γιατί να μην μιλάμε για την προπαγάνδα του ΝΑΤΟ και τις ψεύτικες αποδείξεις που επινόησε η Γερμανία για να δικαιολογήσει τον βομβαρδισμό της Σερβίας και όλη την προπαγάνδα για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο και την οικονομική καταστροφή και τον όλεθρο μιας χώρας και του άμαχου πληθυσμού της να φημώσει την διεθνή μεροληπτική, ιδεολογική, διεθνή δικαιοσύνη για να μην μιλήσει, να, να, να αποσιωπήσει τα μαφιόζικα ψέματα του μαφιόζικου κράτους Κωσυφοπεδίου ε, που ε, για να σώσει το, το εγκληματικό δίκτυο ε, αδιαμέλυσε τη Σερβία. Αυτό είναι ντροπή για έναν αρσατό Ευρωπαίο. Και αντί να κάνουμε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, των Δυτικών Βαλκανίων γέφυρα Ανατολής και Δύσης, τις βάζεται έρμεως στην δυτική επιβολή στην υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η, πολιτική σας για την ένταξη και τη διεύρυνση είναι εμφανώς αντιευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, κυρίε και κύριοι, πρόκειται για μια έκθεση για τη Σερβία. Για... Ο κύριος Επιτιδίος έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια που καταβάλει να γίνει πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω η προσπάθεια αυτή έχει ιδιαίτερη αξία διότι από την σερβία ζητάται να λάβει σκληρέ και σοβαρέ αποφάσει όπω παραδείγματο χάρη να εναρμονίσει την εξωτερική πολιτική τη με εκείνη τη ευρωπαϊκή ενώσεω συμπεριλαμβανομένη και τη ρωσία να μην αποδυναμώσει την αυτονομία ε, τη ε, βοηβοντίνα να χειριστεί εκείνου που έχουν χαρακτηριστεί ω εγκληματίε πολέμου ε, και να αντιμετωπίσει την διαφορετική αντίληψη περί τη ιστορία στην περιοχή. επιπλέον η ενταξιακή πορεία τη έχει συγκυφανθεί με την πρόοδο στι σχέσει με το κωσυφοπαίδιο και την αναγνώριση του κωσυφοπαιδίου που ω γνωστόν αποτελεί το ιστορικό λίκνο του σερβικού ε, έθνου. ενώ όμω από τη σερβία η ευρωπαϊκή ένωση ζητά να είναι συνεπή σε όλε αυτέ τι υποχρεώσει δεν κάνει το ίδιο και με το κωσυφοπαίδιο. εκεί ανέχεται να παραβιάζεται μια βασική αρχή τη δημοκρατία η διάκριση των εξουσιών και η βουλή τη χώρα να ε, καταστρατηγεί και να μην αποδέχεται αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου. δύο μέτρα λοιπόν και δύο σταθμά. οπότε γεννάται το εξή ερώτημα θέλουμε τη σερβία στην ευρωπαϊκή ένωση ή απλώ την εμπέζουμε για να ικανοποιήσουμε τι πολιτικέ επιδιώξει κάποιων κρατών κυρίω τη Γερμανία, που είναι υπεύθυνη για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. ευχαριστώ. και έχουμε ολοκληρώσει τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ακούμε τους ε, ομιλητές με τον κύριο Πρέντα πρώτον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μακάλιστερ για την έκθεσή του που ε, επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Σερβία στην ανταξιακή της πορεία. Χάρη στην πρόοδο αυτή άνοιξαν τα πρώτα διαπραγματευτικά κεφάλαια με τη Σερβία στις 14 Δεκεμβρίου και χαίρομαι ιδιαίτερος για το γεγονός αυτό θα πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην ενταξιακή πορεία της χώρας. Επιπλέον θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση της ρωμανικής μειονότητας. Ο κύριος Μακάλιστερ αφιερώνει μια πολύ σημαντική παράγραφο στην προστασία των μειονοτήτων. Μάλιστα έχω καταθέσει και τροπολογίες για το θέμα αυτό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στα δικαιώματα της ρωμανικής μειονότητας. Θα πρέπει αυτά τα δικαιώματα να γίνουν πραγματικότητα. Πρόσβαση στην ε, ανεξιθρησκεία, στην παιδεία, ε, σε τύπο ε, στην ρουμανική γλώσσα και ούτω καθεξής. Χαιρόμαστε για την εξομάλυση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο, αλλά θα πρέπει να έρθουν περαιτέρω κάποια εμπόδια. Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό Σερβίος, ο κ. Βούτσιτ, θα πρέπει να κάνει μια σαφή επιλογή μεταξύ της ε, θέση της Ρωσίας που είναι υπέρ του προγραμματισμένου ε, δημοψηφίσματος της Ρεπούμπλικα Σέρψκα είναι ευθυγραμμιστή με την ευρωπαϊκή θέση που βλέπει στο δημοψήφισμα αυτό ένα εμπόδιο στην ε, ευρωπαϊκή πορεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Χαίρομαι πάντως για την παρουσία του εκπροσώπου του Συμβουλίου εδώ που στις 15 Φεβρουαρίου θα δεχθεί την υποψηφιότητα για ένταξη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που πιστεύω ότι θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό. Έχετε μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Ξέρετε όμως επειδή θα μιλήσετε μετά δεν μπορώ να σας επιτρέψω. Ο κύριος Φλέκενσταν έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κύριε Μακάλιστερ, αν το αντέχετε άλλη μια έκφραση χαρητηρίων από μένα. Βεβαίω και βλέπουμε ότι πολλά, έχουμε να, πολλά έχουμε, μένουν να γίνουν ακόμη στη Σερβία. Οι πρόοδοι όμως που έχουν επιτευχθεί δεν είναι και αμελητέ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση και με ένα λαό. Σε αυτούς οφείλουμε τι ευχαριστίες για το φιλοευρωπαϊκό πνεύμα με το οποίο έχουν αγωνιστεί όλο αυτόν τον καιρό. Το το Δεκέμβριο του 2015 άνοιξαν τα δύο πρώτα κεφάλαια για τις διαπραγματεύσει. Το κεφάλαιο 35 έχει να κάνει μεταξύ άλλων με την πρόοδο και την εξομάλυνση στις σχέσεις ε, Σερβίας Κοσυφοπεδίου. Βεβαίως και ήταν σωστή επιλογή να ανοίξει ως πρώτο, ένα από τα πρώτα το κεφάλαιο αυτό γιατί είναι εκ να κάνει φόρο εξομάλυνση σχέση σχέση μεταξύ Σερβία και Κωσυφοπεδίου, το να μπορούν τα κράτη αυτή επικοδομητικά να συζητήσουν θέματα περιφερειακή συνεργασία, αλλά και να προχωρήσουν προ ε, προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χέρι-χέρι. Και επίσης, μια και είχε αναφερθεί επαραλημμένως, δεν θα εκπαιδευτώ περισσότερο, αλλά θα σημειώσω και εγώ ότι πρέπει οπωσδήποτε κεφάλαια 23 και 24 να, ξανα, να ανοίξουν ε, όπως άλλωστε επισημαίνει και για τις διαπραγματεύσεις με, με το κοσμοπέδιο η Σερβία, πρέπει πρώτα να ανοίξουν τα κεφάλαια αυτά και να τα τελευταία που θα κλείσουν. Οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να φέρουν πάρα πολύ θετικές εξελίξεις και για την καθημερινή ζωή των πολιτών, γιατί ενισχύουν τη δημοκρατία, ε, εξασφαλίζουν ταχύτατες ε, πρόοδους και προς άλλους τομείς. Αλλά δεν είναι δυνατόν τα κεφάλαια αυτά και οι διατάξεις τους να υλοποιηθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να ε, εμπεδοθούν οι αρχές του κράτους δικαίου με την νομοθεσία. Ε, πρέπει να εξασφαλιστεί μια αλλαγή νοοτροπίας ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως προς τη δικαστική εξουσία και αυτό είναι μια πολιτική που θα πρέπει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως με πιο πολλά κίνητρα και πιο πολλές πιέσεις, περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα τουλάχιστον. Η ε, κυρία Τόμασιτς, παρακαλώ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Έχουν ε, ανοίξει τα πρώτα κεφάλαια στις ε, διαπραγματεύσεις με τη Σερβία και αυτό συνιστά πρόοδο, αλλά δεν θα πρέπει να γελιόμαστε. Δεν έχει λάβει η χώρα κάποια σημαντική καμπή στην σερβική πολιτική. Ε, προσπάθειες τη Σερβίας για σομάλιση το σχέσιο με την Κροατία είναι ελάχιστες. Ε, ακόμη τα θέματα των αγνωμένων ή της αναγνώρισης ύπαρξης στρατοπέδου συγκέντρωσης ε, Κροατών σε σερβικό έδαφος κατά τη διάρκεια του πολέμου της πρώην Οικοσλαβίας, όπως και επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων και των πολιτιστικών αγαθών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και συχνότερα εκπορεύονται πρωτοβουλίε για την κοινή πολιτική άμυνα και τον Ευρωπαϊκό στρατό. Τα κράτη-μέλη όμω και οι πολίτε θα πρέπει να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στου εταίρου και στου γείτονέ του για να αποθέσουν στα χέρια του την κοινή άμυνα. Πώ περιμένετε από του πολίτε τη Κροατία να πιστέψουν στην κοινή πολιτική άμυνα σε μελλοντικού πολέμου, αν ε, μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, κατάφερε να προσπίσει την αξιοπρέπεια των θυμάτων από τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο που έγινε στο ευρωπαϊκό έδαφος εξαιτία πολιτικών συμφερόντων γίνεται όλο και πιο χαλαρή απέναντι στη Σερβία. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κυρία Τόμασιτς, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Σάνι. Έχετε το λόγο κύριε Σάνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Τόμασιτς, φυσικά είστε ελεύθεροι και έχετε δικαίωμα να επικρίνετε ε, ή να ασκείτε κριτική στη Σερβία. Και εγώ μερικές φορές δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με τις μεταρρυθμίσεις ε, στις ε, χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες σταθεροποίησης σύνδεσης. Αλλά πριν από πέντε χρόνια έχει διακοπεί η ενταξιακή διαδικασία. Μήπως εξαιτίας αυτής της διακοπής επιβραδύθηκε και η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Σερβία. Ε, κύριε Σόνι, δεν επιτέθηκε η Κροατία στη Σερβία, αλλά η Σερβία στην Κροατία. Ε, η, Κροατία η, η Σερβία ε, άσκησε επίθεση και έκανε εισβολή. Ενώ ξαφνικά κλείνουμε τα μάτια και είναι σαν να μην συνέβη τίποτα. Τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, τι θα γίνει με τις εκατοντάδες γυναίκες που ήταν θύματα ε, βιασμού και ακόμη ε, δεν αναγνωρίστηκε η δικαιοσύνη για τα εγκλήματα, για τα εγκλήματα αυτά. Δεν είναι λογικό και η Κροατία να αναζητεί ικανοποίηση. Δεν είναι η Σερβία αυτή που θα πρέπει να διεκδικήσει ικανοποίηση. Και Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια οι πολίτες της Σερβίας ε, περιμένουν αγωνίως ε, την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που ξεκίνησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις κυρία Επίτροπε Χράν και ξεκίνησε επιτέλους αυτή η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Έκανε πολλά θετικά βήματα για την περιφερειακή σταθερότητα χώρα αυτή και θα πρέπει να την εκτιμήσουμε, να την αναγνωρίσουμε όπως και η συνεισφορά της ε, στην διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και θα πρέπει να τη στηρίξουμε στους τομείς αυτούς. Θα πρέπει όμως η Σερβία να ε, σεβαστεί τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, όχι μόνο της Κροατικής, αλλά της Βοσνιακής, της Ρουμανικής, επίσης το δικαίωμα σε αυτονομία της Βοηβοδίνας. Όλα αυτά είναι αδιαφυσβήτητα. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ούτε την ανάγκη των δικαστικών μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία, να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια, γιατί χάρη σε αυτό θα γίνει δυνατό δυνατός ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός της Σερβίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, θέλετε μπλε κάρτα ή καρσία. Ε, μα είχατε μιλήσει και νωρίτερα πριν για 1,5 λεπτό είναι αρκετοί οι βουλευτές οι οποίοι θέλουν να εγγραφούν στον κατάλογο για το Καριστιάι. λοιπόν αλλά δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο. Κύριος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς και ισχυρότατου λόγου να υποστηρίζουμε τη διπλή προσχώρηση τη Σερβία. Εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, σημειώνεται σημαντική πρόοδο. Θέλω να συγχαρώ δεν τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση του, η οποία είναι ισορροπημένη στην παρουσίαση των δεδομένων. Ελπίζω να την υποστηρίξουμε όλοι. Για τη, Συρία, για τη Σερβία όμως και ω φίλο τη Σερβίας θέλω να τονίσω κάτι το οποίο υπεγράμμισε και ο αξιότιμος φίλος Charles Τάνακ ότι το κεφάλαιο 30 και κυρίως το 31 του κεκτημένου θα ανοίξει κάποια στιγμή σύντομα. Εγώ ως ιστορικός γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν παραδοσιακές φιλίες μεταξύ των κρατών. Αυτό μπορεί να γύρει ζητήματα γιατί το άρθρο 30 απαιτεί να ανοίξει η πολιτική, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας έναντι ε, παραδοσιακών φίλων Προειδοποιώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί πως καλείται να υπονομεύσει τη σχέση της Σερβίας με παραδοσιακούς τους φίλους στο κεφάλαιο αυτό, γιατί αυτά λένε οι παραδοσιακοί εχθροί της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Φέγα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις επιστρέφω από ε, επίσκεψη στην Κροατία, τη Βοσνία και τη Σερβία. Είναι μεγάλο έθνος ε, η Σερβία, Έναν υπότακτο έθνος, ευρωπαϊκό έθνος. Οι ηγέτες της Σερβίας αγαπούν την Ευρώπη αλλά όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες της Σερβίας θέλουν την Ευρώπη αλλά όχι την Ευρώπη του ριζοσπαστικού Ισλαμισμού όπως ε, εκδηλώνεται στην Βοσνία ή στο Σαντζάκ. Θέλουν την Ευρώπη οι ηγέτες της Σερβίας, την Ευρώπη η οποία σέβεται τους λαούς και τις οντότητες και όχι τα αποσχεστικά κινήματα όπως τη Βοηβοδίνα. Θέλουν μια Ευρώπη χωρίς την κυδαιμονία του ΝΑΤΟ, ή για ηγέτες Σερβίας. Οι ηγέτες Σερβίας θέλουν μια ολοκληρώση ευρωπαϊκή. Οι Σέρβοι όμως δεν θέλουν να μην γίνουν τον, ένα νέο κοσποπαίδιο. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Άρα και το σερβικό... Ε, ε, άρα εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσουμε το σερβικό λαό, το φίλο σερβικό λαό να γίνει Ευρωπαϊκό Λαό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριος Κουκάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια στον Ντέβιτ Μακάλιστερ για την έκθεση που είναι και ισορροπημένη και αντικειμενική. Συγχαρητήρια και στον Επίτροπο Χάν που καθοδηγεί τη Σερβία στις στο, στο αυτών των διαπραγματεύσεων και στον δρόμο που οδηγεί στην ένταξη. Είχαμε ανοίξει κάποια κεφάλαια πέρσι στις διαπραγματεύσει και οι προσδοκίες σε σχέση με αυτή τη χώρα έχουν αυξηθεί. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα για όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή η διαδικασία ολοκλήρωση συνεχίζεται, προχωράει. Η Σερβία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε διάφορες διάφορου τομεί πολιτική. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουμε. Είναι εξίσου ξεκάθαρο, θα πρέπει να ισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί τη χώρα, το κράτο δικαίου και η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, αλλά και οι δραστηριότητε στην περιφερειακή συνεργασία συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου με το κοσυφοπαίδιο. Παρά τη δραματική κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη την περιοχή, ω χώρα που διαπραγματεύεται την προσχώρηση στην Ένωση, η Σερβία χρειάζεται πλουραλιστικά, ελεύθερα ψηλόν, ελεύθερα από πολιτικές πιέσεις. Είναι σημαντικός εταίρος Σερβία στην περιοχή και ένας εταίρος που, στον οποίο θα πρέπει να βασιζόμαστε. Το προσφυγικό έδειξε ότι η Σερβία σε πολλά θέματα ταυτίζεται με τις θέσεις της Ένωσης και είμαι σίγουρος ότι αυτή η στάση θα υπερισχύσει και σε άλλους τομείς εξωτερικής μας πολιτικής μελλοντικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χάουιτ, ο επόμενο ομιλητή, έχετε ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με του υπόλοιπου που χαιρετίζουμε ακριβώ το άνοιγμα αυτό των κεφαλαίων διαπραγμάτευση όπω το 35 για την εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο. Επίση, θα ήθελα το 23 και το 24 κεφαλαίο να ανοίξουν που αφορούν την δικαιοσύνη για όλε τι χώρε υποψηφίε προσχώρηση και το ανέφερα αυτό κυρίω Χάς προηγουμένως. Εδώ έχουμε μια υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε δράση μελλοντική θα πρέπει να αξιολογήσει τη στάση της ε, χώρας μελλοντικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πραγματικά ε, αντιμετωπίζει απειλή έχουμε, η δημοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε 35 επιθέσεις που έχουν καταγραφεί και ένα δίκτυο έχει ε, δημοσιεύσει πληροφορίε ότι τα ανεξάρτητα να θεωρούνται ως κατάσκοποι από τα σκανδαλοφεδερικά έντυπα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε. Και τι γίνεται με τις κοινέ στρατηγικέ ασκήσεις μεταξύ Σερβίας και Ρωσίας. Οι συνάδελφοι σωστά ζητούν αλληλεγγύη ευρωπαϊκή για τη Σερβία μαζί με τα θέματα ασφαλεία, Χαίρομαι όμω που η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει κάποια κονδύλια για τους πρόσφυγες για να βοηθήσει αυτή τη χώρα αναγνωρίζοντας ακριβώς τη δέσμευση της ε, χώρας για την ε, εφαρμογή του, των ποσοστώσεων για τους πρόσφυγες στην Ένωση. Θέλουμε η Σερβία να σε τμήμα των ευρωπαϊκών λύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Μακοβέ, έχετε ένα λεπτό. Η ενσωμάτωση της Σερβίας βεβαίως ε, από μένα γίνεται αποδεκτή αλλά μόνο προς όφελος του πληθυσμού και όχι των πολιτικών της. Πρέπει να σημειώσουμε τα εξή ότι απειλούνται, τρομοκρατούνται από τους πολιτικούς οι δημοσιογράφοι, ακόμη και φυσικές ε, και σωματικές απειλές έχουν δεκτεί. Πρέπει να σταματήσει αυτό για να υπάρχει ανεξάρτητη ε, ανεξάρτητος τύπος. Για τη δικαιοσύνη έχει υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος αλλά πρέπει να υλοποιηθεί και όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εάν δεν υπάρχουν έρευνες, ανακρίσεις και τελικές καταδίκες εις βάρος των λεγόμενων ολιγαρχών επιχειρηματιών που έχουν αποφελθεί τις καταστάσεις. Δεν μπορεί τίποτε να μείνει, να γίνει αξιόπιστο, θα μένουν μόνο σχέδια επιχάρτου και βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί η πρόοδος στον δρόμο της ε, ε, ένταξης. Η Σερβία θα πρέπει να αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική έναντι της Ρωσίας και να ε, στράτευθεί προσυλλομένα προς τη Δύση. Ευχαριστώ πολύ. Ντέλη. Έχετε ένα Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά ο Ντεβιτ Μακάλιστερ έχει τονίσει τα πιο σημαντικά ζητήματα, τα καθοριστική σημασία θέματα για την Σερβία. Από τα όσα μας λέει και η έκθεση πρόοδου έχει προχωρήσει λοιπόν, έχει ανοίξει τα πρώτα και σημαντικά κεφάλαια συνεργάζεται στενά με την Ευρώπη για το μεταναστευτικό και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάντα ξεκάθαρη στο ότι απαιτεί από τη Σερβία η Σερβία έχει κάνει σημαντικές πρόοδους. Πολλά ακόμα μένουν να γίνουν φυσικά για να καλύψει το έδαφος που τη χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη, δημοκρατία, ε, δικαιώματα μειονοτήτων, ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως γιατί η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει τους επόμενους μήνες να κοιτάξουν πολύ προσεκτικά τις πρόοδους στους τομείς αυτούς και να δώσουν το πράσινο φως για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24. Ε, πολλά υποσχόμενα νομοθετήματα και σχέδια δράσης έχουν ε, προωθηθεί αλλά βέβαια κοντός ψαλμός αλληλούι όπως λένε θα πρέπει να υλοποιηθούν κιόλας και θα πρέπει να εξασφαλιστεί κράτος δικαίου στη Σερβία ισοδύναμο και εισάξιο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η ουγγρική μειονότητα μεταξύ της οποίας συγκαταλέγεται και ο υποφαινόμενος πρέπει να χαίρει πλήρων δικαιωμάτων και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η σερβική κυβέρνηση να προχωρήσει στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Και ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τάν. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω εδώ την δέσμευση της Σερβία για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πράγματι συμπεραίνει η Κομισιόν ότι εδώ συγκροτεί ένα μητρό αποτελεσμάτων η Σερβία για την εφαρμογή των κεκτημένων. Και η τακτική της, της Κομισιόν νομίζω έχει αποδώσει καρπούς. Ε, είναι καλό αυτό το μήνυμα έχει κάνει βήματα προόδου η Σερβία για την εξομάλυνση των σχέσεων με, τον, με το Κωσοφοπέδιο και για τη μείωση του προπολογισμού του κρατικού και χαίρομαι τα βλέπω αυτά. Ταυτόχρονα η ανάγκη των διαπραγματεύσεων, το άνοιγμα των κεφαλαίων δεν σημαίνει βεβαίω ότι ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσει και κλείνουν τα κεφάλαια γιατί χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Να τονίσω δύο σημεία. Τον περασμένο Σεπτέμβρη ήμουν στο Gay Parade στο Βελιγράδι και υπήρχε μια ζώνη αστυνομικών που δεν ήταν εκεί για να προστατεύσουν τους συμμετέχοντες στο K Pride ή τον πληθυσμό του Βελιγραδίου κατά τον LGBT. Απλά και μόνο αυτό έδειχνε ότι η θέση αυτών των LGBT είναι πάρα πολύ αδύναμη στην Σερβία. Το δεύτερο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ελευθερία των ΜΕ, το οποίο είναι ουσιοδού σημασία για κάθε δημοκρατία. Είναι επισφαλή η θέση, της, η θέση των ΜΜΕ και έχουμε το Rights ε, που έκανε μια έκθεση και που μιλούσε για την κατάσταση των ε, δημοσιογράφων στη Σερβία. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν πολλή δουλειά ακόμα. να Συγχαίρω τον συντάκτη τον κ. Μακαρίστερ για την ε, εξισορροπημένη δουλειά, αλλά θα ήθελα βεβαίω να δούμε πρόοδο και το άνοιγμα του 23-24 κεφαλαίου ως δείγμα ε, αμοιβές αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε, ε, κύριε Υπουργέ Κούντερ, κύριε Πιτροπεχάνα, κύριε Υπουργέ Γιοξίμοβιτς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ για μία ακόμη αξιόλογη και μεστή έκθεση με θέμα την πρόοδο της Σερβίας ε, και την οποία προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ε, με την κατάθεση τροπολογιών. Ε, χαίρομαι για την έναρξη ε, των, ε, των διαπραγματευτικών κεφαλαίων 31 και 35 για το δημοσιονομικό έλεγχο και την εξομάλυση των σχέσεων με άλλες χώρες, κυρίως με το κοσυφοπαίδιο. Θα πρέπει η ε, Σερβία να, χρησι... να συνεχίσει μεταρρυθμίσει σε δύο συμβατικά κεφάλαια, την ε, δικαστική εξουσία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια. Ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των δικαστών και να εξασφαλιστεί η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ελευθεροτυπία που είναι σημαντικές αρχές και απαραίτητα στοιχεία της ενταξιακής πορείας. Επίσης θα πρέπει να αποπολιτικοποιηθεί η δημόσια διοίκηση και να ε, γίνει περασπίση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων με βάση τις διεθνείς συμφωνίες. Επίσης να εξασφαλιστεί εκπροσώπηση των ε, μειονοτήτων στις διάφορες ε, αρχές τοπικού, περιφερειακού και κεντρικού επίπεδου και πρόσβαση ε, των μειονοτήτων στην παιδεία. Είναι ανησυχητικό ότι με τη ιδιωτικοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σταματούν να εκπέμπουν σε άλλες γλώσσες κάποιοι σταθμοί και επίσης υπάρχει πρόβλημα με τα σχολικά βιβλία. Επίσης θα πρέπει να συνεχιστεί η δίωξη των εγκλημάτων πολέμου σε συνεργασία με το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης για την πρώην ε, Ιουκοσλαβία και επίση ε, να αποφύγουμε το θέμα τη διαβριμένη δικαιοδοσία άλλων χώρων μελών και πίσω με τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά τα θέματα να διαθετηθούν. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Πάβελ, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Μακάλιστερ για την έκθεση του για τη Σερβία και ως πρόεδρος της άτυπης ομάδας Φίλη της Σερβίας και ως Ρουμάνος χαίρομαι για την έναρξη των διαπραγματευτικών κεφαλαίων 32 και 35. Το δεύτερο αφορά την εξομάλυση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο, κάτι που δείχνει τη σοβαρή δέσμευση και αφοσίωση της Σερβίας στην προσπάθεια της ενταξιακής πορείας. Χαιρετίζω και συγχαίρω τη Σερβία για την επικοδομητική της ε, αντίδραση σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική κρίση. Αν συγκρίνουμε την συμπεριφορά της Σερβίας, βλέπω ότι είναι πολύ θετική από τη συμπεριφορά άλλων κρατών μελών. Ε, βέβαια θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ό,τι αφορά την προστασία των μειονοτήτων και τη μη διακριτική μεταχείριση. Επίσης ε, θα πρέπει ε, οι εθνικές αυτές μειονότητε μειονότητες να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, σε ε, διδασκαλία στη μητρική τους γλώσσα και επίσης ε, δικαίωμα στην ανεξαθρησκεία. Πολλές προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν από τη Σερβία και πολλές θυσίες και γι' αυτό θα πρέπει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να στηρίξουν τη χώρα αυτή τις προσπάθειές της, ε, να στηρίξουμε τις προσπάθειες των αρχών και των πολιτών και να δείξουμε ότι η Σερβία έχει πραγματικά τη θέση της στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριο Σπέτερλε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με μεγάλη χαρά καλώς ορίζω τις πρόοδους της Σερβίας όπως τις καταγράφει η έκθεση του συναδελφού Μακάλιστερ. Η έναρξη αυτή των διαπραγματεύσεων συνιστά βήμα προόδου, δείχνει ότι η Σερβία σέβεται τις δεσμεύσεις της. Ελπίζω ότι η Σερβία και μετά τις εκλογές θα τηρήσει την ίδια γραμμή των μεταρρυθμίσεων προς την Ευρώπη. και των καλών σχέσεων με το κοσφοπέδιο. Δεν ε, θα παρασυρθώ σε ε, αγώνα δρόμου με εκείνους που επικρίνουν τη Σερβία. Ελπίζω ότι θα ανοίξει σύντομα το κεφάλαιο 23 και το 24 γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικά για το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον συνάδελφο Μακάλιστερ για την πραγματικά αξιόλογη έκθεσή του για την κατάσταση πρόοδου της Σερβίας το 2015. Το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο με την αναγκαία επακόλουθη αποτελεσματική εφαρμογή, η συμμετοχή σε ειρηνευτικέ αποστολέ, η πρόοδο στην ενταξιακή ε, πορεία τη χώρα αυτή είναι ορισμένα θετικά σημεία. Ταυτόχρονα όμω ε, ε, η έκθεση αναφέρει και ε, κάποιες περσινές ε, πρόοδους ε, που σημαίνει ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της η Σερβία. Η απειλή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η μία παρκώς αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόοδος στο κράτος δικαίου, η συμμετοχή της αντιπολίτευσης σε δημοκρατικές διαδικασίες, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειοψηφιών. Όλα αυτά είναι θέματα που αμελητή θα πρέπει να βελτιώσει η Σερβία. Με το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων σηματοδοτείται η αρχή της θετικής πίεσης προς τη χώρα αυτή για την έναρξη σημαντικών και σοβαρών με, ε, μεταρρυθμίσεων σε μεγάλο αριθμό των μεών. Ε, μένουν όμως ε, σημαντικά θέματα όπως η κρεμότητα σε ό,τι αφορά τους αγνοωμένους, η οριοθέτηση των συνόρων, η κληρονομική διαδοχή, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα της βοηβοδίνας και το καθεξής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Στόκης. Πρόεδρε, ευχαριστώ χαιρετίζω τη διαδικασία αυτή και την έναρξή του στην ουσιαστική τον περασμό Δεκέμβρη. Αλλά για να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο, θα πρέπει κατά τη διάρκεια του τρέχοντο τα κεφάλαια 23 και 24 να ανοίξουν και αυτά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Σερβία θα πρέπει να επιδείξει βούληση και ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις μειονότητες, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει εδώ. Συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων που αναφέρει και η έκθεση του κ. Μακάλιστερ. Παλιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ήταν ιδιαίτερα ελαστική σε σχέση με αυτά τα δικαιώματα και τις χώρες που ήταν υποψήφιες για προσχώρηση. Δεν θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν το ίδιο λάθος με την Σερβία. Ως Ούγκρος από την Ουγγρική κοινότητα ή μειονότητα της ε, Ρουμανίας υποστηρίζω έντονα το θέμα αυτό και έχω υψηλά, ιδιαίτερα υψηλά προσδοκίες όσον αφορά το Μητρό Αποτελεσμάτων της Σερβίας για τα μηνωτικά δικαιώματα. Νομίζω ότι αποτελεί εκ των ΚΑΝΕΦ για την προσχώρηση του χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Λουδίξον. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική. Η Σερβία δηλαδή να προσεγγίσει όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλήσουμε μια νέα φωνή και να στείλουμε ακριβώ αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα, ώστε η Σερβία να αποτελέσει ένα σημαντικό και αξιόπιστο εταίρο. Δέχομαι λοιπόν πολύ θετικά το ψήφισμα αυτό του Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει τι προσπάθειε που έχει ξεκινήσει τι μεταρρυθμιστικέ η Σερβία και που κάνει τα απαραίτητα βήματα για την προσχώρηση στην Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εδώ θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ομοιονοτήτων, των ΜΜΕ, το κράτος δικαίου, δικαιοσύνη. Ίσως τα κριτήρια αυτά να μην υλοποιηθούν άμεσα αύριο, αλλά είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν. Και γι' αυτό ακριβώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Σερβία θα υποστηριχθεί δεόντως γιατί είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε προσέγγιση με τη Σερβία και θα θέλουμε να υλοποιηθεί αυτό σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κολατσέφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Σερβίας εγγυάται την ειρήνη και την ε, ευημερία όχι μόνο για τη Σερβία αλλά για ολόκληρη την περιφέρεια της, για ολόκληρη την περιοχή και έτσι θα πρέπει να ξεπεράσουν τους διχασμούς στην περιοχή. Πολλές είναι οι εθνοτικές ομάδες στη Σερβία, Ούγγροι, Βούλγαροι και πολλοί άλλοι εθνοτικές ομάδες οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν μια ειρηνική συμβίωση. Θα ήθελα επίσης και την παρουσία της ε, Υπουργού των Εξωτερικών να απευθύνω στη Σερβία την έκκληση να επαναφέρει το όνομα του Σάριμπροκ, να εγκαταλείψει το ε, το, το πονίμιο που αναφέρεται σε έναν κομμουνιστή ηγέτη της Σερβίας. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να ερευνούν οι φοιτητές στη μητρική τους γλώσσα. Εάν εξασφαλιστεί και αυτό, θα είναι έτοιμη η Σερβία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε μια μπλε κάρτα, κύριε Κόβατσε, τη δέχεστε. Ζαμπάσκι. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόβατσεφ, συμφωνώ για το Σάριμπροτ και το πονήμιο. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή. Πρώτος στόχος της Σερβίας θα πρέπει να είναι να εγγυάται τις, ε, τα δικαιώματα της βουλγαρικής μειονότητας, να σταματήσει να παρεμβαίνει στο καθημερινό τους βίο, να εξασφαλίζει τα δικαιώματα της βουλγαρικής κοινότητας της Σερβίας. Δεν είναι αυτό μία από τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση της Σερβίας. Απάντηση. Βεβαίως κύριε Τζαμπάσκη είναι προφανώς κύρια προτεραιότητα αυτή και έχει πολύ καλή νομοθεσία για τις εθνοτικές μειονότητες Σερβία αλλά ε, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα βλέπουμε αποστοδρόμηση σε πρακτικές που ανήκουν στο παρελθόν. Βλέπουμε σημάδια ότι είτε σε επίπεδο εισαγγελικών αρχών είτε σε επίπεδο αστυνομικών αρχών ε, υπάρχει δυσμενή μεταχείριση εθνικών, εθνοτικών μειονοτήτων, όπως συμβαίνει με τη βουλγαρική μειονότητα του Σάριμπρο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Βέβαια ξέρετε ότι η μπλε κάρτα ήταν για ερώτηση και όχι για δήλωση είναι προβλέπεται για ερώτηση στην οποία μπορεί μετά να δοθεί ερώτηση. Ο, ο μιλητής είχε πάντω το δικαίωμα να απαντήσει. Κύριε Απόστορα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. στι διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας το πιο σημαντικό ε, θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά θα καταδείξουν πόσο επιτυχημένοι θα είμαστε στην επίτευξη των στόχων μας και στους άλλους τομείς. Υπάρχουν ε, τεράστια κενά ε, στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα διακρίσεων, κυρίως για του ΛΟΑΔ, και η κοινωνία των πολιτών στη Σερβία τη σήμερα ημέρα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να τους υποστηρίξουμε στις δραστηριότητές τους και να φροντίσουμε να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους τομείς πολιτικής που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, βάσει και των αρχών της δημοκρατίας. Ε, υπήρξε μια επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έθεσα το θέμα της ανησυχητικής ε, ε αύξησης της βίας ε, ανδρών κατά γυναικών και ο Πρωθυπουργό μα είπε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η νομοθεσία ώστε να προστατεύονται οι γυναίκε θύματα βία. Ε, πρέπει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα ασφαλεία. Επίση είναι πολύ ανησυχητική η κατάσταση των Ρωμά. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα τη έκθεση. Ε, αναφερόμαστε και στο αντιαθηγανισμό. Διακόπτη πρόεδρο ε, την ομιλήτρια. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Γκουάνο. Μπουονάνο, από τον κύριο Μπουονάνο. Τη δέχεστε. Αρνείται η, η ομιλήτρια. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Πόχε, για ένα λεπτό. Συνάδελφοι, οι σχέσεις ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο πρέπει να αποτελούν ε, ένα από τα κεφάλαια τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει κανεί σήμερα με το κεφάλαιο υπαριθμών 35. Έχω μία ερώτηση για την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξαν διεξοδικότητε συζητήσει ανάμεσα στην κυρία Μογκερίνη και τον ε, πρόεδρο τη κυβέρνηση ε, του Κωσοπεδίου, αλλά δεν ενημερωθήκαμε τίποτα το σημαντικό. Κυρίω το θέμα ήταν ε, το καθεστώς ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, στο Κωσυφοπέδιο. Επίσης, το θέμα της δικαιοσύνης και ρωτώ κατά πόσον έχει απεμπλακεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων και ποιος θα είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι διαπραγματεύσεις. Δέχεστε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Μπονάνο. Όχι και πάλι όχι. Λοιπόν, ε, ξεκίνησε, τέλειωσε ο κατάλογος των αγορητών και ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Κυρία Πέρτη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συνέχιση του ευρωπαϊκού δρόμου της Σερβίας είναι πολύ σημαντικός για την ομαλοποίηση των ε, σχέσεων στην Ανατολική Ευρώπη και ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι ευτυχής για την κατάσταση της Σερβίας κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Γιατί ο στόχος είναι ε, να ελεγχθούν τα μέσα ενημέρωση όρων των μειονοτήτων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να τυπώνται τα κείμενα στα σχολεία στις γλώσσες των μειονοτήτων και αυτό είναι μια σοβαρή παραβίαση ε, της συμφωνίας μεταξύ των κρατών. Ε, ζητώ η Σερβία να αλλάξει την νομοθεσία γιατί η κατ' ουσίαν αποτελεί μία απειλή ε, για την Κροατία και απευθύνομαι στις αρχές της Σερβίας να ξανασκεφτούν ότι το αποκαθεστ... η αποκάθεση του καθεστώτος ε, του 2015 θα πρέπει να επανέλθει, να μην είναι ακραία η πολιτική της Σερβίας, αλλά είμαι σίγουρος ότι η Σερβία θα στείλει σαφές μήνυμα ότι θα σεβαστεί το ε, κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εργαστεί για καλές γειτονικές σχέσεις κοινό στόχος ευρωπαϊκή ένωση και ιδιαίτερα η γερμανία και η αυστρία με την εξωτερική πολιτική που ακολούθησαν κατά τη δεκαετία του 1990 φέρουν σημαντική ευθύνη για τον διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Μετά από μια δεκαετία πολέμων και ανατοϊκών βομβαρδισμών που στόχευαν τη Σερβία, η χώρα αυτή βρέθηκε να έχει απολέσει σημαντικά εδάφη όπου κατοικούσαν σερβικοί πληθυσμοί. Απόλεσε την πρόσβασή της στη θάλασσα, αλλά και το λίκνο του σερβικού πολιτισμού, δηλαδή το Κόσοβο, ενώ σημαντικές υποδομές της καταστράφηκαν σε μια κοινωνία που βρίσκεται έκτοτε σε καθεστώ οικονομική ανασφάλεια, έρχεται η ευρωπαϊκή ένωση και με τον πλέον υποκριτικό τρόπο τη ζητά εδώ και τώρα την απόλυτη προσαρμογή στα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα οργάνωση του κράτου. και σαν να μην έφτανε αυτό η ευρωπαϊκή ένωση ζητά την de facto αναγνώριση του κωσόβου εκ μέρου του βελιγραδίου γεγονό που πέραν των άλλων ενισχύει τον αλβανικό εθνικισμό. επισημαίνουμε το θετικό ρόλο τη Σερβία στο προσφυγικό και δηλώνουμε ότι η θέση της ορθόδοξης σερβίας είναι στην ευρώπη και ο ελληνικός λαός στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της σερβίας. ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντοσιτς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου προς όλους που μίλησαν για ε, την ανάγκη εκδημοκρατισμού της Σερβίας. Αυτό είναι σημαντικό για τα Δυτικά Βαλκάνια συνολικά, αλλά είναι ιδιαίτερα αντιφατική η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ΜΜΕ στη Σερβία, τα οποία αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν να πέσουν όλα στα ίδια χέρια και αυτό θα είναι σοβαρός κίνδυνος για την ελευθερία των μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης. Και ως αποτέλεσμα πολλές μειονοτικές γλώσσες ή καλύτερα μειονοτικά ΜΜΕ που ήταν στις μειονοτικές γλώσσες ε, δεν μπορούν πια να λειτουργήσουν. Αλλά κάθε μειονότητα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται στην γλώσσα της. Αυτό είναι ένα βασικό δημοκρατικό δικαίωμα. Γι' αυτό καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα να παρακολουθήσουν την κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία χρήση όλων των γλωσσών ε, πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Ω εισηγήτρια για το κοσφοπέδιο, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για την συνεργασία που είχαμε τον εισηγητή κ. Μακάλιστερ και να ε, τονίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί μεγάλες πρόοδοι στο διάλογο με το κοσφοπέδιο αλλά και σε άλλα θέματα όπως η καταπολέμηση διαφθοράς κάτι το πολύ σημαντικό επίσης στηρίζω το άνοιγμα δύο κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θέλω η Σερβία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλω και το Κωσφοπέδιο να γίνει μέλος της Ένωσης. Υπάρχουν δύο θέματα που θέλω να θίξω, που με ανησυχούν ιδιαίτερα ως ε, Ευρωπαίο πολίτη. Στο διάλογο μεταξύ Σερβίας και κοσυχοπαιδίου πρέπει να υπάρχει η αρχή της καλής γειτονίας, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι η Σερβία πρέπει να υποστηρίξει την προσπάθεια ένταξη του κοσφοπεδίου στο, στη, για τις ΗΠΑ ή άλλε οργανώσει όπω τη FIFA και την UEFA και όχι να την μπλοκάρει. Γιατί αυτό θα ήταν τμήμα μιας ε, συνεργασία στη διεθνή κοινότητα και θέλω να, καλήσω, να καλέσω τι αρχέ τη Σερβίας να μην στέλνουν τα δικαιώματα ορισμένων ε, επικριτικών δημοσιογράφων γιατί αυτό είναι μέλος της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Καφτάλντο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου Μακάλιστερ περιλαμβάνει αρκετά σημαντικά θέματα με τα οποία συμφωνούμε. Το πρόβλημα του δικαστικού συστήματος που ακόμα ε, καθυστερεί και υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις. Η διαφθορά ε, ένα φαινόμενο το οποίο επιμένει και φυσικά υπάρχει και η διάκριση κατά των ε, ευάλωτων ομάδων, τους ΛΟΑΔ και τις γλωσσικές μειονότητες η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης ε, στην πολιτική διαδικασία και να μην αναφερθώ και στην ε, πολύ ακόμα στρατιωτική ρητορία. Ε, αυτή τη στιγμή όμω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κακό. Υπάρχει το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία. Γιατί επιμένουμε να το θεωρούμε αυτό ω πρόσκομα και, ως, και όχι ω ένα εργαλείο για να ξαναξεκινήσουμε εμεί έναν ειλικρινή ε, πολιτικό διάλογο και να θέσουμε επιτάπητο στα ζητήματα τα οποία μας διέρεσαν στο παρελθόν. Διότι και οι δικέ μας οι πολιτικές είναι πολύ αμφίσιμες και ποικίλουν. Από τη μια ζητάμε ε, να... Ε, υπάρχει ακαμψία και από την άλλη ζητάμε διαπραγμάτευση για το Nord Stream. Θα πρέπει λοιπόν να επικρατήσει η λογική για να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μπορεί και να μην επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάλτσο. Ευχαριστώ πολύ. την έκθεση για τη Σερβία θα ήθελα να αναφερθώ στη θέση των γλωσσικών μειονοτήτων. Δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα ε, η νομοθεσία όπως ε, ζήτησε το Συνταγματικό Δικαστήριο. Υπήρχε καταληκτική προθεσμία για το τέλος του 2014. Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε ε, να εγκριθεί η σχετική νομοθεσία το στομότερο δυνατόν. Τα εθνικά συμβούλια έχουν χάσει τις περισσότερες από τις εξουσίες τους, δεν είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, έχουν ε, αλλάξει άρδιν, δεν υπάρχουν μειονοτικές γλώσσες στον προγραμματισμό των καναλιών και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά από τη σερβική ε, κυβέρνηση να εφαρμόσει διεθνείς συμβάσεις. Αλλά δεν αρκεί αυτή η έκκληση. Οι διεθνείς συμβάσεις ε, πρέπει να εφαρμοστούν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και πιο στεναρή διατύπωση η οποία θα ζητά από τη Σερβία να τις εφαρμόσει. Η κυρία Σούικα, καταρχάς, Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μακάλιστερ για τη θαυμάσια έκθεσή του που περιέχει όλα τα θέματα που συζητήσαμε τα τελευταία χρόνια αλλά με τις πολλές τροπολογίες ε, που συμπεριέλαβε από εμάς τους Κροάτες που βοηθούν το κείμενο. Αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες από προηγούμενες εκθέσεις που αναλαμβάνουν εδώ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν έχουν γίνει πολλά και πρέπει να γίνουν πολλά από την Σερβία. Η εξωτερική πολιτική της Σερβίας πρέπει να συμβαδίζει με την αντίστοιχη της Ένωσης. Ιδιαίτερα το βήμα την, για τη σχέση με τη Ρωσία. Και εφόσον ε, ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει αυτό το δημοψήφισμα στην ε, Σερβική Δημοκρατία, θα είμαστε πάντα αντίθετοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν θέματα με την αυτονομία της Βοηβοντίνα και την αναγνώριση της πολιτιστικής πολυμορφίας, καθώς και η τύχη των αγνωμένων. Θα επιμείνουμε από αυτού, αλλά είμαι πεπισμένη ότι θα επιλύσουμε διμερώς τα προβλήματά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούγορ. Ευχαριστώ πολύ. Τα πρόσφατα βήματα στις σχέσεις Σερβίας-Ένωσης έχουν προκαλέσει μια επιτάχυση της πορείας προς την ε, ένταξη. Αυτό είναι καλό. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να τονίσω πώς έχει η κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα. Κατά την ε, διαδικασία ενταξιακών διαδικασιών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμό ο οποίος θα δώσει αναφέρετα δικαιώματα στον πληθυσμό της Βοηβοντίνα και θα ενισχύσει τα εθνικά συμβούλια και θα ρυθμίσει όλους τους τομείς πολιτικής που θεωρούνται σημαντικοί από τις αναγνωρισμένες οργανώσεις των ε, μειονοτήτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η πείρα έχει καταδείξει ότι μετά την ένταξη μιας χώρας πολύ συχνά υπαναχωρούν για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως ακριβώς συνέβη στη Ρουμανία και τη Σλοβακία μετά την ένταξη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και εκτιμένα, πριν την ένταξη στη Ρουμανία, για παράδειγμα το 2005, είχε κριθεί ένας νόμος για τις μειονότητες, αλλά τώρα μετά την ένταξη δεν έχει εφαρμοστεί τελειωτικά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τελευταία ομιλήτρια από τον κύριο Μπλόκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να συγχαρώ τον Σάλφο Μακάλιστερ για αυτή την πολύ ενθαρρυντική έκθεση. Η Σερβία έχει σημειώσει σημαντικές προόδους και στις 14 παρελθόντος Δεκεμβρίου ε, ανοίξαμε τα κεφάλαια 31 και 35 η Σερβία απέδειξε λοιπόν ότι είναι αξιόπιστος ε, εταίρος στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η κίνηση των προσφύγων που διασχίζουν τη Σερβία συνεχίζεται. Είναι λοιπόν αναγκαίο να διασφαλίσουμε ένα ε, θετικό μέλλον για τις επόμενες γενναίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τη Σερβία να εφαρμόσει οικονομικές μεταρρυθμίσεις με την προενταξιακή βοήθεια για να τις επιτρέψει να βελτιώσει τις υποδομές της και μετά τα κεφάλαια 24 και 25 επίσης πρέπει να βοηθήσουν για τη μεταρρύθμιση στο δικαστικό κλάδο γιατί υπάρχουν δυσχέρειες στους τομείς αυτούς ωστόσο ο εκδημοκρατισμός της ε, σερβικής κοινωνίας είναι προϋπόθεση για να οδεύσουμε προς την ε, επιτυχία και την ευημερία της Σερβίας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι λίγη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής της Προέδρου. Επόμενος ομιλητής είναι ο Επίτροπος κύριος Χάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία αντικατοπτρίζει και πόσο σημαντική είναι η διαδικασία της διεύρυνσης, διότι πρόκειται για έναν σταθεροποιητικό παράγοντα ε, κομβική σημασίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την περιοχή. Ε, σαφώς χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να ξεπεράσουμε το κληροδότημα του παρελθόντος και όπως είπα και στην εισαγωγή μου θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα διμερεί ζητήματα δεν θα παρακολύσουν τη διαδικασία προσχώρησης αλλά η διαδικασία της ε, ε, συμμόρφωσης είναι μια πολύ σημαντική ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση με τη Ρωσία δεν αποστέλει το σωστό μήνυμα υπ' αυτήν την έννοια. Η αποτελεσματική και αμερόληπτη αντιμετώπιση εγκλημάτων πολέμου αποτελεί μία από τις πολύ σημαντικές προτεραιότητές μας στις διαπραγματεύσεις με τη Σερβία. Θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή των μέτρων που έχει ε, προβλέψει η Σερβία στο πρόγραμμα δράσης της, στο κεφάλαιο 23, για την ανάγκη για αποτελεσματική και αμερόληπτη μεταχείριση σε θέματα εγκλημάτων πολέμου ε, ίση μεταχείριση υπόπτων, ε, ποινές και προστασία των θυμάτων. Επίσης, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας το θέμα της προστασίας των εθνικών μειονοτήτων. Αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη Σερβία το θέμα αυτό. υπάρχει η προεργασία και παρακολουθούμε στενά την συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη τη Σερβία, κυρίως σε θέματα παιδείας, χρήση γλωσσών και πρόσβαση θρησκευτικές υπηρεσίες και μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μειονοτικές γλώσσες. Η Σερβία πρέπει να διασφαλίσει βέβαια στην πράξη την διασφάλιση όλων αυτών των δικαιωμάτων. Και πάλι θα παρακολουθούμε λοιπόν κατά πόσο επικεντρώνεται η Σερβία στην εφαρμογή των μέτρων που ανέλαβε βάσει των προγραμμάτων δράσης της για το κράτο δικαίου και το σχετικό πρόγραμμα δράσης για τις εθνικές μειονότητες. Και πάλι θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη έκθεση. Ευχαριστώ εκείνους που συνεισέφεραν στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό Κούντερς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έκθεση και για τη δέσμηση του εισηγητή, του κυρίου Μακάλιστερ έχω την εντύπωση ότι ε, η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Η Σερβία έχει κάνει ένα θετικό βήμα, κυρίως στον τομέα του κράτους δικαίου και την εξομάλυση των ε, σχέσεών της με το Κωσυφοπαίδιο. Κύριε Μακάλιστερ, αναφερθήκατε στην ανάγκη να ε, ανοίξουν τα κεφάλαια 23 και 24. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να σας πω ότι βάσει αυτής της νέας προσέγγισης, το... οι κανόνες στα κεφάλαια 23 και 24 είναι ε, το θέμα το οποίο θα εξετάσουμε αρκετά νωρί. Βέβαια πρέπει να γίνει και η σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει η προεργασία στι σχετικές ομάδες εργασίας για να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό και κάποιοι θα ήθελαν να, βλέπουν, να ακούσουν και μεγαλύτερη πρόοδο για τι εθνικέ ε, μειονότητε. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης το οποίο παρουσιάζεται σήμερα από τη σερβική κυβέρνηση και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχει διάθεση για την επίλυση των διμερών προβλημάτων. Στα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου του το Συμβούλιο καλεί τη Σερβία να εντατικοποιήσει την διαδικασία μεταρρυθμίσεών της ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ανέφεραν και αρκετοί από εσά σήμερα. Δικαστικό σώμα, καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο. Επίση, κάποιοι από εσά ανέφεραν και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να γίνεται πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων, ιδίω ε, των Ρωμά, καθώ επίση και την αποτελεσματική εφαρμογή τη νομοθεσία για την προστασία των μειονοτήτων. Ε, με ε, βάση και τη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή φυλετική ταυτότητα και φυσικά βελτιώσεις ε, στο περιβάλλον και στο επενδυτικό κλίμα. Επίσης, ε, κάποιοι επέκριναν την ε, ελευθερία του λόγου και του τύπου. Σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και σε αυτά τα θέματα και νομίζω ότι ο κύριος Χάν αναφέρθηκε και στην ενεργό αντιμετώπιση των, προ... των εγκλημάτων πολέμου. Θα πρέπει επίση η Σερβία να προχωρήσει τη διαδικασία εξομάλυση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο που είναι ένα από τα καθόδη ζητήματα και νομίζω ότι υπήρξε σημαντική πρόεδρο από πλευρά ε, Σερβίας ε, προσέγγισε το Κωσυφοπαίδιο και νομίζω ότι θα το θίξουμε αυτό και στη συζήτηση για το Κωσυφοπαίδιο αργότερα. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν και στην εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την ευθυγράμμιση των ε, υποψήφιων χωρών με τι ε, εξωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχέση με τη Ρωσία και σύμφωνα με την ε, τελευταία έκθεση Προέδρου, Προόδου Είχαμε 65% ευθυγράμμιση και πρέπει η Σερβία σιγά σιγά να ευθυγραμμίσει τις πολιτικές της με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας και αυτά θα εξεταστεί στα πλαίσια του κεφαλαίου 31. Όπως γνωρίζουμε η Σερβία δεν ε, ε, συμμορφώθηκε, ε, μάλλον δεν ακολούθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στις κυρώσεις προς τη Ρωσία και το 2015 υπήρχε και το θέμα της Προεδρίας του ΩΣΑ. Ελπίζουμε να υπάρξει και ευθυγράμμιση στο θέμα αυτό στο μέλλον. Βάσει και της νέας μας προσέγγιση, τα κεφαλαία 23 και 24 για το κρέτος δικαίου θα συζητηθούν αρκετά νωρίς στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που ε, αποστέλει και ο εισηγητής και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω λάβει ένα σχέδιο ψηφίσματος. Κλείνει η συζήτηση.